Hi everybody. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, όσοι θέλουν να παραμείνουν σε αυτό το συναρπαστικό πάνελ που θα ξεκινήσει τότε, να καθίσουν στις θέσεις τους. Όλοι, όσοι θέλουν να συνεχίσουν τις συζητήσεις, να εξέλθουν παρακαλώ από την αίθουσα, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω. Δεν φταίμε εμείς. Ε, τα προηγούμενα πάνελ καθυστέρησαν. Έχουμε ένα καταπληκτικό πάνελ πολύ ψηλού επίπεδου και είναι κρίμα να τους στερούμε χρόνο με περαιτέρω καθυστέρηση. Wow, silence in the room. Great. Ωραία ησυχία στην αίθουσα, λαμπρά. Αλλά θα περιμένω λίγο ακόμη. Ready to go. Great. This ώσπου να φύγουν όσοι δεν ενδιαφέρονται. Το πάρελ μας θα ασχοληθεί με την καινοτομία στο τουρισμό και την ψηφιακή οικονομία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχουμε για να δούμε πώς θα σπαστούμε την ψηφιακή επανάσταση, την καινοτομία, τις πλατφόρμες για να ωφελήσουμε έναν από τον πιο αραγδαία ανερχόμενο κλάδο τη Ευρωπαϊκή οικονομία, τον τουρισμό. Και ευχαριστώ θερμότατα τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οργάνωση αυτή, γιατί πραγματικά θα πρέπει να φέρουμε τον τουρισμό ω κλάδο ε, που είναι κλειδί τη οικονομία μα και κινητήριο μοχλό θέσεων απασχόληση ε, στο επίκεντρο του προγράμματό μα. Γιατί χάρη στον τουρισμό θα αναζωογονηθεί η Ήπεθρος, ε, οι πιο απόμακρε περιφέρειε, θα εντάξουμε καλύτερα στι κοινωνίε του μετανάστε μα. Χρειαζόμαστε θέσεις απασχόλησης και ελαστικές θέσεις απασχόλησης και για τους νέους μας. Εγώ είμαι Ιταλίδα, παρόλο που εκλέγομαι στη Σουηδία και βλέπω πως ε, τη τρέλα έχουν οι Σουηδοί για την Ιταλία, αλλά βλέπω ότι και οι Ιταλοί αρχίζουν ε, και τρελαίνονται για τη Σουηδία. Και μάλιστα η οικογένειά μου έχει μια τουριστική επιχείρηση στην Ευρώπη. Είναι μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, οπότε γνωρίζω ε, πολλά από τα προβλήματα, τις προκλήσεις ε, τους πονοκεφάλους ε, των επιχειρήσεων αυτών με το TripAdvisor, το Booking.com, την Amazon και πώς έχει να αλλάξει όλα αυτά, όλες αυτές οι εξελίξεις, τον τρόπο λειτουργίας τέτοιων επιχειρήσεων. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την αγαπητή φίλη Μαρία και Επίτροπο Μαρία Γκαμπριέλ. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρουμε την μεγάλη σας δέσμευση για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία χρόνια ολόκληρα και τώρα είστε εδώ ως Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τα θέματα αυτά. Επίσης έχουμε κοντά μας και τον Υπουργό Τουρισμού της Ρουμανίας, τον κύριο Ντόμπρε, την κυρία Μοντέρα Ντεγκιάρ, Ευρωβουλευτή, μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον αγαπητό συνάδελφο Νίκολα Ντάντι, που είστε, α, ε, από κοινού διαχειριζόμαστε το την έκθεση για την ε, ε, οικονομία ε, και τη οικονομία της συνεργασίας. Επίσης έχουμε τον κύριο Πατανέ, τον καλωσορίζουμε θερμά και την κυρία Σανταντέρ που είναι εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών και τον κύριο Λάιρβακ που είναι αντιπρόεδρος για βιομηχανικά ζητήματα και εταιρική ευθύνη του, της ομάδας IT Αμαντέους και τον κύριο Χελδράν, που είναι Υπουργό Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος της Μούρσια την κυρία Ντανιέλη που είναι καθηγήτρια οικονομικής πολιτικής και διευθυντρία του Master of ε, Οικονομίας και Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Βοκόνη τον κύριο Φερχόβεν, τον Γενικό Διευθυντή και Διαχειριστικό Διευθυντή της Booking.com και τον κύριο Καρμπαντέλα που είναι πρόεδρος της Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εταιρείας Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόθεση του τουρισμού. Ε, θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις πολλαπλές προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιακή επανάσταση και πώς επηρεάζει αυτή τον τουρισμό που έχει επιφέρει ρηξικέλευτες αλλαγές και επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις και τις πτυχές του τουρισμού. Επίση, να αποτίσω φόρο τιμή στους καταπληκτικούς μας επιχειρηματίες ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί αυτοί πρωτοστατούν στον κλάδο και εμεί, ε, ω πολιτικοί θύνοντες ε, ε, νιώθουμε μεγάλη ταπεινοφροσύνη, γιατί δεν είμαστε πια εμείς ηγέτες. Εμείς θέλουμε απλώς να διευκολύνουμε, και αυτό είναι το καθήκον μας, να διευκολύνουμε, να χειραφετήσουμε, να ενδυναμώσουμε, να διαμορφώνουμε τα νομικά πλαίσια που θα εξασφαλίζουν μια ασφάλεια δικαίου, θα είναι στεγανά ως προς τις μελλοντικές εξελίξεις, θα είναι ουδέτερα από άποψη διαδικτύου και θα βοηθούν στην αξιοποίηση των τεράστιων επιχειρηματικών δυνατοτήτων. Όλα αλλάζουν. Ο τρόπος που κάνουμε κράτηση των πτήσεών μας, που κάνουμε κράτηση για τις διακοπές μας, ο τρόπος που πληρώνουμε για όλα αυτά και φυσικά και οι μεταφορές. Όλα αλλάζουν. Και θα ξεκινήσω με μια βόμβα που θα ρίξω. Θα ταράξω τα νερά το θέμα των δεδομένων, γιατί εδώ ασχολούμαστε και με την οδηγία για την ιδιωτικότητα στο, στο διαδίκτυο, την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα που μας έχει δημιουργήσει τεράστιο πονοκέφαλο και να το συνδυάσω με τις δυνατότητες ανάπτυξης και καινοτομία του τουρισμού, γιατί είμαστε μια οικονομία που, που επικεντρώνεται στα δεδομένα. Ο τουρισμός σίγουρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό και αν στο μέλλον κάποιος πράκτορας θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα, τα mail, τη διάθεση mail, τον, ε, τα, τηλέφωνα των πελατών σας για να τους στέλνει μια προσφορά τα Χριστούγεννα, θα πρέπει να ζητούμε την συγκατάθεση του πελάτη εκ των προτέρων για να τον βάλουμε στη βάση δεδομένων. Χρειάζονται για όλα αυτά ρυθμίσεις, κανονιστικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν και την, τον τουριστικό κλάδο. Και γι' αυτό περιμένω τις απόψεις και να σας πω ότι προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της προσωπικής ακεραιότητας, της ιδιωτικότητας, της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας και της ε, ε, προσπάθειας να μην επιβραδύνουμε την εσωτερική ψηφιακή αγορά και να μην επέβουμε σε αυτή, κάτι που είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι αντικρώμενα μερικές φορές τα συμφέροντα. Έχουμε δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις, μία για τις πλατφόρμες τις επιγραμμικές, τις προκλήσεις ε, και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα γύρουμε τείχους απέναντι σε τρίτες χώρες και ε, επιτυχής πολυεθνικές και το πώς θα ε, διαθέτουν τα προϊόντα τους, αν θα τις κατηγορούμε, θα τις δαιμονοποιούμε ή θα άρουμε τα δημοκρατικά εμπόδια και τους φραγμούς στη γραφειοκρατία και τον υπερβολικό κανονιστικό πλαίσιο που έχουμε στην Ευρώπη, ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για να μπορέσουν και οι ευρωπαϊκές εταιρείες να ανθίσουν και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, να γίνουν πρωταθλήτριες και αυτές Νίκολα, εσύ θα μας πεις για τη μάχη που δίνουμε για τη συνεργάσιμη οικονομία, συνεργατική μάλλον οικονομία και ε, να δούμε τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, επιχειρήσεων πελατών και ούτω καθεξής, γιατί όλα αυτά έχουν αλλάξει και οι παραδοσιακοί τελεστές αντιμετωπίζουν πολλέ προκλήσει έω και απειλέ μερικέ φορέ. Θα πρέπει να του βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν τι δυνατότητε τη συνεργατική οικονομία, λειτουργώντα στο σωστό πλαίσιο, φορολογία, αγορά εργασία, ασφάλειες, ε, ε, ευθύνε, υποχρεώσει. είναι εθνικά θέματα. Εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι μπορούμε να κάνουμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο εν συντομία για την αρχή, στην αγαπητή φίλη και πάλι, την Επίτροπο Μαρία Γκαμπριέλ, και ελπίζω ότι θα έχουμε ζωηρή συζήτηση μετά. Θα προβλέψουμε κάποιο χρόνο και για τη συζήτηση. Μαρία, εσύ πρώτη για 7 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Άννα Μαρία, αγαπητή Πρόεδροι, ε, Υπουργοί, συγγνώμη, Ευρωβουλευτές. Ε, ευχαριστώ καταρχήν θερμά τον Πρόεδρο Ταγιάννη για την εξαιρετική ε, και πολύ επίκαιρη πρωτοβουλία γιατί μιλάμε για την οικονομική, για την ψηφιακή επανάσταση που βιώνουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας. Οπότε το να απομονώσουμε τον τουρισμό από την ε, ψηφιακή αυτή επανάσταση ήταν το λάθος. Ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω το όραμά μου, κάποιες από τις ιδέες μου, αφενός και αφετέρου, να παρακολουθήσω με ενδιαφέρον τις δικές σας παρατηρήσεις, να ακούσω τις δικές σας εμπειρίες. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά να ε, αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση, δηλαδή να έχουμε μια συζήτηση όπου ο τουρισμός θα συναντήσει την ψηφιακή οικονομία και θα επωφεληθούν και οι δύο κλάδοι, αμοιβαία. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε με το διάλογο, με τη συνεννόηση, αλλά και με την κοινή μας επιθυμία να υλοποιήσουμε τους κοινούς στόχους, γιατί δεν μπορούμε να αποφεύγουμε τέτοιες συζητήσεις τις οποίες ανταμώνουν ο τουρισμός και ο ψηφιακός κόσμος, γιατί η, η ψηφιακή οικονομία αγγίζει όλους τους κλάδους. Έχει ενταχθεί στην καθημερινότητά μας. Και αν θέλουμε να ανθίσει ο ευρωπαϊκός τουρισμός, ε, και να φτάσουν το ωφέλη του σε όλους τους πολίτες, δεν μπορούμε να ξεχνούμε τις νέες τεχνολογίες. Το διαδίκτυο, διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο, ζωτικό στόχο στον τομέα των ταξιδιών στην Ευρώπη και το επιγραμμικό περιεχόμενο είναι η πρωταρχική πηγή πληροφοριών για τα ταξίδια και ξεπερνάει όλες τις άλλες μορφές των συμβατικών μέσων ή του παραδοσιακού μάρκετινγκ στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, οι αυτοματοποιημένες σχέσεις με τον πελάτη, οι κρατήσεις που γίνονται online, το checking που γίνεται επίσης online. στατιστικά το online περιεχόμενο είναι το 40 υπεύθυνο για το 49% τουριστικών αφήξεων στην Ευρώπη. Βέβαια, θα πρέπει να πάρουμε κάποια απόσταση και να δούμε ποιε είναι οι συνέπειε αυτών των αλλαγών. Θα πρέπει να το υπενθυμίσουμε ότι ο τουρισμό ε, αντιπροσωπεύει το 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και 5,2% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού περίπου, δηλαδή 10 εκατομμύρια θέσει εργασία. Επίση, είναι η Ευρώπη ο πρώτο τουριστικό προορισμό παγκοσμίω, με 600 περίπου εκατομμύρια τουριστικέ αφήξει το χρόνο. Πώ λοιπόν το διαδίκτυο και ο ψηφιακό κόσμο ή βάλει αυτή την κόσμος συμβάλλει σε αυτή την δυναμική ε, οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει καταρχήν η ψηφιακή οικονομία να εξυπηρετεί τον τουρισμό. Θα πρέπει να έχουμε κοινού κανόνες ώστε να καταπολεμούμε τα εμπόδια και τους φραγμούς για τα αγαθά που προσφέρονται. Επίσης, η εξελίξη στον βιογραφικό αποκλεισμό θα επιτρέψει σε όλους τους καταναλωτές να αγοράζουν το διαδίκτυο τα αγαπημένα τους προϊόντα ε, όπου και αν διαμένουν ή όπου και ταξιδεύουν και να μπορούν να, ε, να λαμβάνουν στα στις χώρες που ταξιδεύουν τα προϊόντα με τους ίδιους όρους που θα τα παραλάμβαναν και στην πατρίδα τους. Θα Ήθελα να σας αναφέρω μερικά θέματα που μου είναι ιδιαίτερα προσφύλη. Καταρχήν, χαίρομαι που καταργήθηκα τα τέλη περιαγωγή. Ας μην το ξεχνούμε. Έχουν περάσει μόλις τρεις μήνες από την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Αλλά έτσι ο κόσμος που θέλει να κρατήσει τις επαφές με τους οικείους του, αλλά και να χρησιμοποιήσει στον επαγγελματικό βίο τα θέματα αυτά. Χθε είδαμε από το Ευρωβαρόμετρο ότι το 72% των Ευρωπαίων γνωρίζουν τους νέους κανόνες για την περιαγωγή και μάλιστα άρχισαν ήδη να αλλάζουν τις συνήθειές τους. Σε μερικές χώρες η αύξηση της χρήσης των δεδομένων είναι εξαπλάσια σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε μας λένε όλες οι ενδείξεις ότι μερικοί παροχοί μετά το τέλος των τελών περιαγωγής επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δικτύωση στι τουριστικέ ζώνε χάρη στην αύξηση τη ζήτηση που οφείλεται στην κατάργηση των τελών περιαγωγή. Ένα άλλο σχέδιο που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ είναι το σχέδιο Wi-Fi για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Wi-Fi for EU. Έτσι δίνουμε πρόσβαση στους ταξιδιώτες στην Ευρώπη ε, σε ένα δίκτυο που θα έχει 8.000 σημεία επαφής ακόμη και σε χωριά της Ευρώπης. Γιατί αν έχουμε κάτι που πραγματικά είναι ιδιάζον και εξαιρετικό είναι ότι καταρχήν για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει άμεση επέμβαση στις τοπικές κοινότητες και δεύτερον από τη στιγμή που ε, κάνει login κανείς εγγραφή σε ένα σημείο ταυτόχρονα εγγράφεται και στα 8.000 σημεία που υπάρχουν ανά την Ευρώπη. Οπότε δεν χρειάζεται να ξαναγραφεί μετά. Πρόκειται επίση για μια πρωτοβουλία που αφορά το περιεχόμενο. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη περισσότερων και καλύτερων ψηφιακών υπηρεσιών από του ε, τοπικού παρόχου. Ηλεκτρονικό τουρισμό, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι καλή υποψήφη. Επίση, ε, και τα τουριστικά θέματα περνάνε σε ε, επιγραμμική διάσταση. Και μέχρι στιγμής ένα μικρό αριθμό των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό εμπόριο για να συνδεθεί με του ε, ε, ε, δυνητικού πελάτε. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει και θα συμβάλλει και ο τουρισμό στην αλλαγή αυτή. Για παράδειγμα, κάποιε προκατακτικέ αναλύσει μπορούν να βοηθήσουν τα ξενοδοχεία να προσωποποιήσουν τι επιχειρήσει του, να τι εξατομικεύσουν και να προσφέρουν στοχευμένε προσφορέ για αναβάθμιση ή για συμπληρωματικέ υπηρεσίε πώς εξηγείται αυτή η ανισορροπία. Η απάντηση δυστυχώς είναι απλούστατη. Ε, έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων. Πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν έχουν την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή ικανότητα να επενδύσουν στις ψηφιακές τεχνολογίες. Οπότε είναι εύλογες οι ανησυχίες τους για το πώς αυτό επηρεάζει το επίπεδο απασχόλησης, τις συνθήκες απασχόλησης και τον επιμερισμό των κερδών ή των εισοδημάτων. Σήμερα η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών στον τουρισμό ε, απαιτεί νέες δεξιότητες, ώστε όλοι οι τελεστές του κλάδου να γίνουν ε, ε οι κύριοι της μοίρας τους και των αλλαγών αυτών. Θα πρέπει επίσης να καθησυχάσουμε του πολίτες και να δημιουργήσουμε πρόσφορο έδαφος, ώστε η μετάβαση προς την ψηφιακή οικονομία να είναι υποφελής και για τους καταναλωτές σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να αυξήσουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την επιμόρφωση και την κατάρτιση για να βελτιώσουμε την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Δεν σας αναφέρω πολλά στοιχεία. Μόνο το 37% του ενεργού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βασικές στοιχειώδεις ψηφιακές δεξιότητες. Ενώ ξέρουμε ότι από το 2020 το 90% των θέσεων απασχόλησης θα απαιτούν τέτοιες ψηφιακές δεξιότητες. Βλέπετε λοιπόν τι χάσμα δημιουργείται και καλούμαστε να το γεφυρώσουμε. Και ο κλάδος του τουρισμού ίσως επηρεαστεί περισσότερο από όλου, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και βασικός μοχλός και κινητήριο δύναμη και να πρωτοστατήσει στις εξελίξεις. Και γι' αυτό θα ήθελα να απευθύνω έκκληση για να διαμορφωθούν εθνικές συμμαχίε που δεν θα είναι από σήμερα πια 17 αλλά 18 γιατί ε, έχει προσχωρήσει και η Σλοβακία. Θέλω λοιπόν όλες οι χώρες να ενδύνουν τις προσπάθειές τους, γιατί όλοι όσοι βρίσκεστε εδώ γνωρίζετε ότι οι εθνικές συμμαχίες για τις ε, ψηφιακές θέσεις απασχόλησης είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να προωθήσει την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και να αφουγκραστούμε τις ανάγκες κλάδων όπως του τουρισμού για να ανταποκριθούμε πιο άμεσα στις προκλήσεις τους. Θα με ρωτήσετε πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε νέες αγορές υπηρεσιών. Η απάντηση είναι η ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα πρέπει όμως να προωθήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και την διαλειτουργικότητα. Κάτι τέτοιο θα μα επιτρέπει να αναπτύξουμε καινοτόμε υπηρεσίε για να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει του τουρισμού να αξιοποιήσουν το ανεκμετάλλευτο δυναμικό του. Επίση, κάτι τέτοιο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Αυτές οι επιγραμμικές πλατφόρμες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον κλάδο και χρησιμοποιούνται κυρίως για τις κρατήσεις, το μάρκετινγκ, τη σχέση με τους πελάτες. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες όπως το Expedia, το Booking.com, το TripAdvisor είναι έτοιμα της καθημερινότητάς μας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα υγιές οικοσύστημα όπου θα σκείται θεμητός ανταγωνισμός από όλους τους οικονομικούς φορείς και οι άδικες πρακτικές δεν θα ε, επιδρούν ε, στους καταναλωτές. Αυτό θα το πούμε και στην ενδιάμεση αξιολόγηση και στις αρχές του επόμενου έτους θα υποβάλουμε νομοθετική πρόταση για να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τέτοιου είδους αθέμητες πρακτικές που κυρίως πλήττουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον τουρισμό. Γιατί στον τουρισμό έχουμε πολλές επιχειρήσεις και πολλούς ανθρώπους που υφίστανται τις δυσμενείς συνέπειες αυτών των αθέμητων πρακτικών. Επίσης, ε, η, η ψηφιακή κουλτούρα είναι πολύ σημαντική για τις ε, επιλογές των ε, ταξιδιών. Και μάλιστα 45% των ε, ερευνών που γίνονται για τουριστικούς προορισμούς γίνονται μέσω του διαδικτύου. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την παρουσία φορέων που προωθούν ε, την πολιτιστική κληρονομιά, γιατί τέτοιος πολιτιστικός τουρισμός ε, ε, σημειώνει άνοδο. Για παράδειγμα, το Rijksmuseum του Άμστερνταμ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο των, στις, στους πίνακες και παρόλα αυτά δεν έχει μειωθεί ο αριθμός των επισκεπτών, εξακολουθεί να είναι το Rex Museum, τα πιο πολύ συχνά στα μουσεία του κόσμου. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα στην Ιταλία, την Ισπανία. Έχουμε το Europeana. Επιμένω γιατί δεν χρησιμοποιούμε παρκώ αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Είναι σημαντικό λοιπόν υπάρχουν τέτοια σχέδια που θα επιτρέπουν στους τουρίστες χάρη στην τεχνολογία να έχουν περισσότερες προσφορές, γνώσεις και έτσι να προσφέρουμε και στον κλάδο περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη έχει απαράμιλο δυναμικό για να προσελκύσει τουρίστες από όλο τον κόσμο και η ψηφιακή οικονομία θα μπορέσει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο και να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον θεμητού ανταγωνισμού κυρίως ε, για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του τουρισμού ώστε να καταρρύψουμε όσο περισσότερους φραγμός γίνεται και να διευκολύνουμε την απρόσκοπτη κυκλοφορία ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών που έχουν κέρια σημασία και για τον τουρισμό. Και ελπίζω να έχουμε τακτικά διάλογο ώστε να αναλάβουμε αυτή την κοινή προσπάθεια για να έχουμε μια, ένα μοναδικό τουριστικό κλάδο στην Ευρώπη, ανταγωνιστικό, πλήρη ευκαιριών και ε, ευθυγραμμισμένο με την ψηφιακή επανάσταση. Ε, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε γιατί βλέπω διαφορά. Τότε που ήμουν Ευρωβουλευτής μου κόβατε το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ που τώρα με αφήσατε να μιλήσω μέχρι τέλους. Ποτέ δεν θα σε διέκοπτα Μαρία γιατί αυτά που λες είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ε, ως Επίτροπος κυρία Γκαμπριέλ μπορείτε να βασιστείτε στην συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εφαρμόσουμε όλα αυτά για τα οποία μας μιλήσατε και περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία το θεματολόγιο για τις ψηφιακές δεξιότητες. Μεγάλη τιμή είναι τώρα για μένα και μεγάλη χαρά να έχω εκ δεξιών μου τον Υπουργό Τουρισμού της Ρουμανίας, κύριο Τίτους Ντόμπρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να παραστώ σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή, ειδικά για τη Ρουμανία. Θα πρέπει να είναι και σημαντική στιγμή για την Ευρώπη, πιστεύω. Ε, ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Ταγιάννη, διότι τον ενδιαφέρει ο τουρισμός και ανέκαθεν τον ενδιαφέρε. Παρακολούθησα τις δηλώσεις του με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η τεχνολογία και η καινοτομία έχουν αλλάξει σημαντικά τις συνήθειες των τουριστών και αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση που οφείλει κανείς να κάνει και να τη λάβει υπόψη του. Τα τελευταία 25 χρόνια ε, διαπιστώνουμε ότι η τεχνολογία συνεχώς αναπτύσσεται, αυξάνεται, εξελίσσεται. Στην Ρουμανία η αύξησή της ήταν ε, εκθετική. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη ως προς τη ταχύτητα των μεταφορών των δεδομένων και αυτό είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα μου οι τουρίστες και όχι μόνο οι τουρίστες αλλά και οι πολίτες ενημερώνονται καλύτερα με ε, την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων και έτσι προωθούνται νέα επιχειρηματικά πρότυπα στον χώρο του τουρισμού. Η νέα ψηφιακή οικονομία είναι εδώ και πρέπει να την προσαρμόσουμε αλλά και να προσαρμοστούμε σε αυτήν για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Ο δημόσιος τομέας αλλά και ο ιδιωτικός τομέας οφείλουν αμφότεροι να μπορούν να, εκπληρώσουν τα προαπαιτούμενα της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι ψηφιακές πλατφόρμες μας επιτρέπουν να προωθήσουμε καλύτερα τους προορισμούς και να προσφέρουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να στραφεί στον τουρισμό, να κινηθεί προς τον τουρισμό σε αυτό το νέο ε, πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο. Ο τουρισμός είναι μια πολυσχηδής ε, δραστηριότητα και γι' αυτό εδώ γίνεται λόγος και τα κύριο λόγο για την Ευρώπη. Και όπως και άλλοι το υπογράμμισαν, πράγματι η Ευρώπη είναι ο υπαριθμόν ένα τουριστικός προορισμός παγκοσμίως και ακριβώς λόγω αυτού, αυτής της πρωτιάς οφείλουμε να παίρνουμε τον τουρισμό πολύ σοβαρά υπόψη. Οφείλουμε να ε, κάνουμε σοβαρό διάλογο για τις επενδύσεις τις τουριστικές, επενδύσεις ιδιωτικής προέλευσης. Οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι ο τουρισμός είναι ένα πεδίο δόξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ο κλάδος που δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την ευκαιρία να αναπτυχθούν εφόσον έχουν ένα έξυπνο ανεπτυξιακό και επιχειρηματικό σχέδιο και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κλάδο του τουρισμού να έχει ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, για να στηρίξει ε, τις υποδομές και τις υπηρεσίες. Πράγματι η Ευρώπη είναι ο ένα τουριστικός προορισμός παγκοσμίω. Ο αριθμός των τουριστών που έρχονται στην Ευρώπη συνεχώς αυξάνει και χρειαζόμαστε εκτεταμένες υποδομές για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ροές. Το πρόγραμμά μας πρέπει να είναι συνεκτικό, να έχει συνοχή, συνέπεια και να ε, συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωσή του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνεργατική οικονομία κομίζει προστιθέμενη αξία και για τους καταναλωτές και για τους επιχειρηματίες ευκαιρίες και συμβάλλει ε, ταυτόχρονα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην επίτευξη της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αναπτυχθεί η συνεργατική οικονομία με υπεύθυνο και νόμιμο τρόπο, σύνομο μάλλον τρόπο. Ε, και γι' αυτό οι πολιτικές για την οικονομία διαμοιρασμού θα πρέπει να ρυθμιστούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε παιχνίδι επί ίσης όρες. Δεν πρέπει να ε, δημιουργήσουμε ιδιαίτερους και ειδικού κανόνες για ορισμένες επιχειρήσεις ή για ορισμένους σχηματισμούς. Αντιθέτως, οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύσουν στους ε, πάντες, σε όλους. Και θα πρέπει να ρυθμίσουμε και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Να σας δώσω λίγα παραδείγματα και δεν θα αναφερθώ καθόλου ονομαστικά. Έχουμε πλατφόρμες που είναι δραστήριες στη ρουμανική αγορά που δεν έχουν ε, ε, ρουμανικό αφημί, δεν έχουν καταχωριστεί ε, στη, για λόγους φορολογίας. Έχουμε μια πλατφόρμα μόνο που έχει καταχωριστεί την ΕΞ, η οποία πληρώνει κανονικά τους φόρους της σύμφωνα με την ρουμανική νομοθεσία. Ας πούμε ότι υπάρχει εταιρεία αυτή η οποία λέγεται Χ. Και έχουμε τώρα μια άλλη πλατφόρμα, ψη να την πούμε, που δεν έχει καταχωριστεί, δεν έχει ρουμανικό αφημί, δεν εκδίδει αποδείξεις ε, ε που να ισχύουν ε, στην, ε, στις ρουμανικές αρχές, αλλά, αλλά δραστηριοποιείται εντός Ρουμανίας αλλά και εκτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι υποχρεωμένη να ε, καταχωριστεί ως πάροχος τουριστικών υπηρεσιών εντός της Ρουμανικής επικράτειας, διότι λέει ότι παρέχει αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν. Όπως γνωρίζετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζουμε να μην έχουμε ευρωπαϊκό μοντέλο εγγυήσεων για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Πρέπει να μιλήσουμε για τις διαδικτυακές συναλλαγές το Ρουμανικό κράτος, το ε, Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Τουρισμού έχουν νομοθετήσει για να ρυθμίσουν ε, για την παροχή υπηρεσιών ε, βραχυπρόθεσμης διαμονής. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα γιατί η βραχυπρόθεσμη διαμονή το μόνο που κάνει είναι να αυξάνεται, να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Η ενοικίαση δηλαδή βραχυπρόθεσμης διαμονής. στη Ρουμανία γίνεται συζήτηση στη δημόσια σφαίρα για ένα σύστημα τεχνολογίας και πληροφοριών που θα ανοιχνεύει και θα καταγράφει τις τουριστικές δραστηριότητες. Μία νέα νομοθεσία η οποία θα αρχίσει να ισχύει από Πρώτου του 2018 προβλέπει τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων συλλογής, ανάλυσης, διάδοσης, συγκέντρωσης δεδομένων και διαμόρφωση σχετικών δικτών για τις τουριστικές ε, δράσεις και δραστηριότητες. Νομοθετούμε λοιπόν και ρυθμίζουμε το τοπίο ε, της ανάλυσης όλων αυτών των δεδομένων. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα το διαχειριστεί αυτό το σχέδιο ε, το Υπουργείο Τουρισμού και οι, Εθνικές υπηρεσίε ε, Υπηρεσίες ε, Επικοινωνιών. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων θα γίνει πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο οι πάροχοι των τουριστικών υπηρεσιών υποχρεούνται να συλλέγουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα για όταν κάνει check-in ο τουρίστας και αρχής γενομένης αυτών των δεδομένων που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των τουριστών, όχι μόνο αυτών που είναι στην Ρουμανία αλλά και των τουριστών που έρχονται από το εξωτερικό, θα μπορέσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα. Όλα αυτά γίνονται προς όφελος της ασφάλειας και θα ήθελα να μιλήσω και για τον έξυπνο τουρισμό τον ευφυή τουρισμό. Θέλουμε μια ευφυή προσέγγιση ε, γιατί όλοι μπορούν να αξιοποιήσουν και να ωφεληθούν από τις ευφυείς στρατηγικές. Ε, οι εστιατόρες, τα καταλήμματα, ούτω καθεξής. Όταν έχουμε έξυπνα συστήματα, συστήματα μεταφορών, ε, ίδρευσης, ε, επικοινωνίας εντός των πόλεων, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μειώνεται το κόστος. Έχουμε την Άλβα Γιούλια, μια πόλη στη Ρουμανία, στο κέντρο της περιοχής της Τρανσιλβανίας. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά η Τρανσιλβανία το 2016 κηρύχθηκε ο υπεριθμόν ένα ε, τουριστικός προορισμός παγκοσμίω από τον ταξιδιωτικό οδηγό Lonely Planet. Και ε, η συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και τοπικών ε, αρχών ήταν πραγματικά αγαστή και μπορέσαμε να αναπτύξουμε αυτό το πρόγραμμα για τις έξυπνες πόλεις στο εξωτερικό. Όλα αυτά εντάχθηκαν στη στρατηγική ανάπτυξη ανάπτυξης 2014-2020 σε συνεργασία και σε συνεργεία και με την Παγκόσμια Τράπεζα. Τα ωφέλη ήταν πολύ σημαντικά εμείς θα έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωση το πρώτο εξάμεινο του 2019 και αυτό είναι και ευθύνη αλλά και ευκαιρία. Είναι ε, ευκαιρία έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τον τουρισμό να αποκτήσουν συνέργεια. Ε, είναι πράγματι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που θα στηρίξει την ενθάρρυνση του τουρισμού, θα στηρίξει τα ταξίδια, θα προστατεύσει τους καταναλωτές και θα εξασφαλίσει την ασφάλεια. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε, ε, κύριε Υπουργέ. Ε, περιμένουμε με ανυπομονησία να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη Ρουμανία, να επισκεφθούμε και πάλι αυτή την ε, χώρα και θα σας ευχαριστώ που τονίσατε τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το λόγο έχει η Κλαούδια Μοντέρο Αγγιλάρα από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 4 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άννα Μαρία. Καταρχήν, να μην ξεχάσουμε την ε, Παγκόσμια Μέρα του Τουρισμού που γιορτάζουμε σήμερα και να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έθεσε τον τουρισμό, το σημαντικό αυτό κλάδο, στο επίκεντρο του προγράμματός μας και διοργάνωσε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Ο παγκόσμιος ε, τουρισμός ε, διακινεί κάθε χρόνο 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπου. Επίσης, μέχρι το 2020 οι μετακινήσει των τουριστών θα φτάσουν στο 1,8 δισεκατομμύρια. Με βάση τα στοιχεία του Ιανουαρίου του 2017 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τουρισμού στην Ευρώπη μπήκαν 620 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή 50% ε, των ε, διεθνών αφήξεων. Ε, Επίσης, δεδομένου του ο τουρισμός είναι μιας, ένας κλάδος που ανέρχεται, είναι το 48% των, της εξαγωγής υπηρεσιών στην Πορτογαλία, είναι ένας τομέας που ε, αφορά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται. Επίσης, είναι κατακόρυφος ε, και πολυσχηδής ε, και πολυδιάστατος. Πρόκειται για ένα προϊόν που δίνει ο τουρισμός που είναι τόσο σημαντικό για την Ευρώπη και τον κόσμο που έχουμε την ε, ανάγκη και το καθήκον να το προστατεύσουμε ενώ απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες του. Επίσης, έχουμε τη, τον κόσμο της ψηφιοποίησης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας. Ε, θα πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη στον Στον τουρισμό η ζήτηση είναι ελαστική και η προσφορά όταν είναι ακαμπτή δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη ζήτηση που ακολουθεί κάποιες τάσεις και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Σήμερα έχουμε ένα πιο κατατοπισμένο τουρίστα, πιο απαιτητικό, που θέλει ε, αυθεντικές εμπειρίες, εξατομικευμένες, ε, θέλει να έχει στα χέρια του τη μοίρα του και να συμβάλλει στην ε, αυτοανάπτυξη και αυτοεκπλήρωσή του η καλύτερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στις ρηξικέλευτες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα έχει ένα όνομα και το όνομα αυτό είναι καινοτομία. Η καινοτομία και η βελτίωση είναι απαραίτητε να βελτιώσουμε την κατάσταση, να καινοτομήσουμε και να είμαστε καλύτεροι από τους ανταγωνιστές. Και φυσικά θα πρέπει να διατρέξουμε κάποιους κινδύνους για να τα κάνουμε όλα αυτά. Και αυτή είναι η πρόκληση του κλάδου. Ε, και δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στη στήριξη των νεοφιών επιχειρήσεων του τουρισμού. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και να συμπαρασταθούμε στις υπάρχουσες επιχειρήσεις, να δώσουμε ε, να, διευκολύνουμε στη διαφοροποίηση της προσφοράς ε, και στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, να προωθήσουμε ε, κλάδους και προϊόντα ε, ιδιαίτερα μικρής ζήτησης και να λάβουμε υπόψη και την τεχνολογία και φυσικά τον σημαντικό ρόλο των νέων που έχουν την τεχνογνωσία, έχουν τις δεξιότητες, έχουν τα προσόντα που είναι πιο ενημερωμένα, προσαρμοσμένα στις εξελίξεις. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες και χώρο στους νέους να προσαρμόσουν το παραδοσιακό στο σύγχρονο. Ο τουρισμός αξίζει και κάποια συγκεκριμένα μέσα και μηχανισμούς από την Ένωση που θα προσαρμόζονται στις νέες επιχειρήσεις, στους νέους επιχειρηματίες και θα συνδυάζει τη δημιουργία πλούτου και δημιουργία θέσεων απασχόληση με την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισορροπιών. Χρειάζονται κίνητρα, συγκεκριμένες ε, δημοσιονομικές ε, γραμμές και στήριξη. Ελπίζω στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο να έχουμε ειδική δημοσιονομική γραμμή για τον τουρισμό, όπω ε, ζητήθηκε επανειλημμένω. Έχει νόημα μια κοινή πολιτική τουρισμού. Επίση, να μην ξεχνούμε την ανάγκη τη καινοτομία, προσαρμογή στην ψηφιακή οικονομία, την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και την προώθηση, τη, τη διαφοροποιημένη προώθηση μέσω των διαφόρων πλατφορμών. Και πέραν των αναγκών που έχει ο τουρισμός, χρειάζεται περισσότερο αναγνώριση και υποστήριξη από χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Και τέλος να αναφέρω δύο πράγματα για την ψηφιακή οικονομία. Ε, χρειαζόμαστε νέες πλατφόρμους κινητικότητας και στέγασης. Έχουμε την δημιουργία έξυπνων προορισμών και έξυπνων προϊόντων. Εδώ και τρία χρόνια μιλούμε για τους περιορισμούς και τις προκλήσεις και τις αλλαγές που χρειάζονται για τις ε, πλατφόρμες κινητικότητας. Χρειαζόμαστε πιο άμεση δράση και πιο συνεχή δράση. Θα πρέπει, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει το διαδίκτυο των πραγμάτων να το λάβουμε υπόψη μαζί με τα παραδοσιακά προϊόντα για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη μόχλευση για την οικονομία και επίσης να επιτρέψουμε δημιουργία αξίας, ε, πλούτου και απασχόληση στον τουρισμό. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και σίγουρα ο τουρισμός ε, αξίζει την υποστήριξή μας και την προσήλωσή μας για να μπορέσουμε χάρη σε αυτό να δημιουργήσουμε μόχλευση για την οικονομία των περιφερειών μας και της Ευρώπης ολόκληρης πάρα πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αγαπημένο μου φίλο, τον κύριο Ντάντη, ο οποίο είναι μέλο τη Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και Προστασία Καταναλωτών και ήταν επίση και εισηγητή τη έκθεση για την ε, συνεργατική οικονομία. Νίκολα, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε τέσσερα λεπτά να εκφράσω τις απόψεις μας. Ε, η έκθεσή μας ε, προϋπόθεσε, προϋπέθεσε πολύ μεγάλη δουλειά. Βεβαίως ε, θέλω να πιστεύω ότι ο τουρισμός έχει υποφεληθεί από την ε, ψηφιακή επανάσταση. Η συνεργατική οικονομία έχει λάβει ένα σημαντικό μια σημαντική όθεση από την ψηφιοποίηση. Υπάρχουν πλέον πολλές ευκαιρίες, πολύ περισσότερες, γιατί έχει διαφοροποιηθεί η τουριστική προσφορά. Υπάρχουν πλατφόρμες ε, ε, που ε, προσφέρουν πολλές δυνατότητες της φιλοξενίας, δηλαδή υπάρχουν και νέες επαναστατικές μέθοδοι τουριστικής προσφοράς. Εμείς έχουμε καταθέσει μια έκθεση μετά από την δήλωση της Επιτροπής, γιατί είναι προφανές ότι η συνεργατική οικονομία ε, σίγουρα με πολλά πλονεκτήματα έφερε όμως και κάποια ανισορροπία στα παραδοσιακά συστήματα. Είναι σαφές ότι οι ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα η συνεργατική οικονομία στον τουριστικό τομέα είναι πάρα πολλές. Έχουμε τη διαφοροποίηση της προσφοράς, πολύ σημαντική. Από την άλλη βέβαια, στην αγορά εμφανίζονται πολλές ε, τουριστικές ευκαιρίες ε, σε μέρη που ήταν ε, περιφερειοποιημένα, που δεν είχαν αξία με τα παραδοσιακά κριτήρια. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτές οι πλατφόρμες συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Ε, δεν θέλω τώρα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά έχουμε σήμερα ε, πολλούς ενδιαφέροντες νέους προορισμούς για τουρισμό. Με όλες, ή ε, όλες αυτές τις ευκαιρίες τις αναλύσαμε και μαζί και τους κινδύνους. Γιατί στον κίνδυνο υπάρχουν βεβαίω νέες δυνατότητες, αυτές έχουν αλλάξει την τουριστική προσφορά, και ως εκ τούτου είναι σαφές ότι υπάρχουν και νέες δυσκολίες κυρίως διότι η τουριστική αγορά μέσα και από τις πλατφόρμες εκτίθεται και σε άτομα που δεν είναι επαγγελματίες. Είναι οικογένειες οι οποίες έχουν ε, τη δυνατότητα να νοικιάσουν τα σπίτια τους, τα διαμερισματά τους, ε, τα ε, δωμάτια τους, ακόμα και τα κρεβάτια τους. Και έτσι λοιπόν η... θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές ε, νομικό πλαίσιο που να διαχωρίζει τον επαγγελματία από τον μη επαγγελματία και να είναι ξεκάθαρα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για τους επαγγελματίες είναι σαφές ότι θα πρέπει να, υπάρχει η ίδια, να υπάρχουν οι ίδιες δυνατότητες πρόσβασης. Για τους ερασιτέχνες και εκεί τα πράγματα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα για να μην υπάρχει παράνομη και αθέμητος μάλλον ανταγωνισμός. Εξάλλου, να είναι σαφή και τα δικαιώματα των τελικών χρηστών. Και αυτό πολύ σημαντικό. Γιατί χρησιμοποιούν ε, δομές που δεν είναι επαγγελματικές. Κατόπιν και το θέμα που έθιξε και η Επίτροπος ε, στην παρέμβασή της, το θέμα των πλατφορμών ε, εκεί όπου γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών για την προσφορά και τη ζήτηση, αυτό είναι λάθος. Εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε μόνο τις ε, πλατφόρμες εκείνες που είναι σε άμεση σχέση με τις τοπικές αρχές. Χρειαζόμαστε ε, πλατφόρμες οι οποίες θα ε, συνοδεύονται και από κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις, από κάποια μορφή φορολογίας. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε σε αυτόν τον τομέα, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, πρέπει να έχουμε πλατφόρμες ε, που αποδίδουν φόρους, από τις οποίες προκύπτει εισόδημα. Αυτό που συμβαίνει με πολλές πλατφόρμες σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη είναι ότι τελικά προκύπτουν παρατυπίες ε, και τελειώνω γιατί νομίζω ότι δεν έχω πια χρόνο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι σήμερα η συνεργατική οικονομία ρυθμίζεται περισσότερο από τα δικαστήρια και λιγότερο από τα κοινοβούλια. Εγώ θεωρώ ότι κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να χαράξει ένα απλό νομικό πλαίσιο όπου θα είναι όμως και σαφές ποιες είναι οι υποχρεώσεις των παρόχων, επαγγελματιών και μη, ποια είναι τα δικαιώματα των χρηστών και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των πλατφορμών. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία και με άλλους ε, θεσμούς. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε πολύ που η θέση μας είναι σχεδόν κοινή ε, με μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε για τις ε, πλατφόρμες. Το Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει τη δουλειά πάνω σε αυτό και βεβαίως ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά. Επόμενη η κυρία Αντωνιώνη, η οποία είναι καθηγήτρια στο Μποκόνι, στο Μιλάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κύρια Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος κύριος Ταγιάννη μας εξήγησε τα τεκτενόμενα στον τουρισμό, μίλησε για την τεχνολογία, για την ανταγωνιστικότητα, ε, βεβαίως και κάτω από το πρίσμα της παραγωγικότητας. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα πράγματα που αναφέρθηκαν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διαβεβαίωσω όλους, γιατί εγώ περισσότερο ασχολούμαι με την επιστήμη και την έρευνα, να διαβεβαιώσω λοιπόν όλους ότι ε, ο τουρισμός θα πάει πάρα πολύ καλά και θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και λόγω της ε, τεχνολογίας. Η τεχνολογία ήταν και παλαιότερα εκείνη η οποία επέτρεπε να κάνουμε κάποιες ε, κρατήσεις. Το 80, 80 υπήρξε ήδη μια τεχνολογική πρόοδος ε, έγινε κάποια οριζόντια αλλά και κάθετη εξέλιξη. Το 2000 φτάσαμε στο διαδίκτυο και αυτό οδήγησε και σε μείωση των τιμών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη διαμεσολάβηση. Νέες μορφές ε, κρατήσεων. Ε, κλείνω λοιπόν αυτή την ιστορική αναδρομή γιατί θέλω κυρίως να ασχοληθώ με το θέμα της ε, sharing economy, της συνεργατικής οικονομίας όπως αναφέρεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, και κάτι για την οικονομική πραγματικότητα, ε, κάποια στοιχεία για τα ρομπότ, γιατί νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ε, δώσει μια κατεύθυνση τι θα γίνει ε, τελικά με όλους αυτούς που θα εκδιωχθούν λόγω της ε, μεγαλύτερης εμφάνισης ε, των ρομπότ. Για την εικονική πραγματικότητα θέλω να πω ότι σήμερα δεν ακούσαμε και πάρα πολλά, δεν ακούσαμε να γίνεται λόγος για αυτή την εικονική πραγματικότητα. Ε, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, κυρίως ε, και στα μουσεία και σε χώρους ε, που στον τομέα του πολιτισμού μπορεί κανείς να κάνει πολλές και νέες εμπειρίες. Άρα και αυτό είναι κάτι το σημαντικό. Ας επανέλθουμε όμως ε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συνεργατική οικονομία, στις ε, πλατφόρμες. Είπαμε προηγουμένως ότι η συνεργασία πρέπει να υπάρχει, αλλά με μια τελείως νέα μορφή. Ε, και πού θα σταματήσουμε. Ε, πλέον έχουμε από τη Wikipedia που φτάνουμε μέχρι πάρα πολλά άλλα, πολλές ειδικέ περιπτώσεις. το Uber μεταξύ μας δεν πέφτει κιόλα σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει το Airbnb, αυτό ναι, το επίπεδο της πλατφόρμας. Όλα αυτά έχουν ε, προσελκύσει πάρα πολλές επενδύσεις και με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αν θέλετε είναι μία μικρή αγορά που σιγά σιγά επεκτείνεται, διευρύνεται αλλά μην ξεχνάμε ότι ε, σε ένα πραγματικό χρόνο και σε παγκόσμια κλίμακα το να μπορεί κανείς να κάνει πράγματα αυτό αλλάζει πάρα πολλά και δεν κοστίζει κιόλα. Είναι εργαλεία που κοστίζουν όλο και λιγότερο, μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει και με το κινητό του. Ε, βασίζονται βέβαια στην εμπιστοσύνη. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο υπάρχει η τυραννική δημοκρατία της ζήτησης ε, όπως ε, χαρακτηριστικά αναφέρεται. Έχουν προκύψει ε, αλλαγές σε μια έντονη συζήτηση για το ότι όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Τώρα, για την συνεργατική οικονομία, το 16 στην έρευνα, των 28, το 50% των καταναλωτών γνώριζαν τις πλατφόρμες της ε, συνεργατικής οικονομίας, αλλά μόνο το 17% ε, χρησιμοποιεί και στην ίδια έρευνα, αν δούμε λιγάκι τους νέους μέχρι 39 ετών, ε, το 32% χρησιμοποιεί αυτές τις πλατφόρμες, που σημαίνει ότι μέσα σε λίγο μόνο χρόνια αυτοί οι άνθρωποι ε, θα μεγαλώσουν ηλικιακά. Ως εκ τούτου θα υπάρξουν πάρα πολλές δυνατότητες χρήσης ε, των πλατφορμών. Και μόνον αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Το 2013 μιλάγαμε για 10 δις ευρώ και για το 2020 Μιλάμε για 500 δις ευρώ. Μία, ένας κλάδος που αναπτύσσεται πολύ περισσότερο από την παγκόσμια οικονομία και αυτό, αυτά τα στοιχεία έχουν σχέση με τα ξενοδοχεία, με τις επιχειρήσεις, βεβαίως και με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, για να ξέρουμε έτσι λιγάκι το τι ακριβώς διαδραματίζεται. Ε, βλέπω ότι δεν έχω πια άλλο χρόνο, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο-τρία θέματα. Τέσσερα λεπτά είχατε. Λοιπόν, εάν η ζήτηση είναι ιδιαίτερα ενεργή, τότε και η προσφορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται με τις πλατφόρμες, να δώσουμε όμως τη δυνατότητα και στις τοπικές αρχές να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να εκφράσω. Το δεύτερο είναι αφορά στη διαφάνεια. Μιλήσαμε για, την, για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Νομίζω ότι στο Ταλίν ελέγχθησαν κάποια θέματα για το web tax. Ε, περιμένουμε να υπάρξει μια συμφωνία σε ευρύτερη κλίμακα, σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό που έχει σημασία και θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα είναι το θέμα της εργασίας. Γιατί εμείς ε, ε ασχολούμεθα με την αγορά εργασίας και βλέπουμε ότι ενώ ε, πολλοί φεύγουν από τον παραδοσιακό τουρισμό, οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερη τεχνολογική πρόοδο, οι επιχειρήσεις εκείνες είναι που προσφέρουν θέσεις εργασίες. Σε αυτήν μπορεί κανείς να βρει απασχόληση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσον αφορά το θέμα της ε, ε, τεχνητής νοημοσύνης, κατά την άποψή μου, ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την τεχνητή αυτή νοημοσύνη η οποία όμως στον τουρισμό που έχει ένα τεράστιο δυναμικό ε, μπορεί να βοηθήσει. Το θέμα είναι ότι στην Ευρώπη το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς ε, οι οποίοι φεύγουν από τον τουρισμό. Έχουμε την ε, οικονομία, την συνεργατική, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει και νέες θέσεις απασχόλησης. Θα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε ε, με την ε, επιστημονική σας κατάρτιση και τώρα θα ήθελα να περάσω στον κύριο Λούκα Παντανέ. Για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ όλους. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και σε σχέση με όσους άκουσα σήμερα εγώ ασχολούμαι με τον τουρισμό και τελικά την, τη ζωή μου ε, και οι γονεί μου και οι προγενέστεροι αυτών έζησαν στον τουρισμό. Ελπίζω το ίδιο να συμβεί και με τα παιδιά μου. Αυτό που ενδιαφέρει σήμερα είναι να δούμε τι μπορεί να προσφέρει ο τουρισμός ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ελέγχθηκαν σήμερα πάρα πολλά πράγματα και πολλά από αυτά που θα ήθελα να πω εγώ τα είπαν ήδη άλλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, θα πω κάποια πράγματα που είναι σημαντικά. Υπάρχει το θέμα των big data. Αυτό το μελετώ εδώ και κάποια χρόνια, γιατί προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ε, στις επιχειρήσεις του κλάδου μας. Σήμερα το πρόβλημα είναι ότι ε, θα πρέπει κανείς ε, να γνωρίζει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν να εξοικειωθούμε καλύτερα με τους πελάτες μας, με τους τουρίστες. Ο πρόεδρος κύριος Ταγιάννη ανέφερε κάποια στοιχεία για τον τουρισμό και εμείς ε, να πούμε το εξής. Ξέρουμε πόσοι έρχονται, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ε, πόσα δαπανούν οι τουρίστες. Έτσι μπορούμε κατά προσέγγιση να πούμε, αλλά δεν ξέρουμε πόσα ακριβώς δαπανούν και πόσα θα μπορούσαν να δαπανήσουν. Άρα δηλαδή είναι σημαντικό να μην εξετάζουμε μόνο τον αριθμό των τουριστών, αλλά κυρίως στο πόσα δαπανούν και πόσα θα μπορούσαν να δαπανήσουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η ποιότητα, όχι μόνο η ποσότητα. Ε, το να γνωρίζουμε καλύτερα τον τουρίστα αυτό σημαίνει, παραδείγματο χάρη, ένας ε, Κινέζος μπορεί να έρθει στην ε, Ευρώπη να ε, κάνει εδώ τουρισμό, αυτός ο Κινέζος μπορεί να έρθει τουλάχιστον 10 φορές στην Ευρώπη. Και αυτές τις 10 φορές θα πρέπει όμως να βιώνει κάτι διαφορετικό, να έχει μια διαφορετική τουριστική εμπειρία. Σήμερα έγινε επανειλημμένα λόγος για την αηφορία. Στην ε, Ευρώπη, η Ιταλία έχει πάρα πολλά ιστορικά κέντρα, κέντρα μεσαιωνικά κέντρα και ως εκ τούτου ε, μπορεί κανείς να προσφέρει μια πλούσια τουριστική εμπειρία. Ακριβώς αυτό που ε, επιθυμεί η ζήτηση. Και εμείς αυτό κάνουμε. Η χρήση της ε, πλατφόρμας, κατά την άποψή μου, αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, για να είναι ανταγωνιστικές, για να μπορέσουν να επιβιώσουν στην κρίση. Σήμερα ζούμε μια στιγμή πολύ σημαντική για μας. Δηλαδή, ε, πλέον μπορεί κανείς να γνωρίζει καλύτερα το τι απαιτείται και να προσαρμόσει αυτό την προσφορά του. Η πλατφόρμα όσον αφορά στην, στις διάφορες πλατφόρμες που υπάρχουν πολλά εξαρτώνται και από το γεγονός ότι η αγορά μας είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη και πολλές φορές ε, δεν υπάρχει θάρρος εκ μέρους των αρμόδιων αρχών για να λάβουν και τις σχετικές αποφάσεις. Ε, παραδείγματος, αν υπάρξει ο φόρος αυτός ε, στο το περίφημο web tax, αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι επωφελήθηκαν, μπόρεσαν να αναπτυχθούν και σήμερα μάλιστα έχουν και κυρίαρχη ε, θέση στην αγορά. Είναι δύσκολο να ε, ανταγωνιστεί αυτούς τους ε, μεγάλους παίκτες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάρα πολλές ευκαιρίες έχουν κλείσει. Κατά την άποψή μου λοιπόν σε αυτό το θέμα του WebTax υπάρχει ουσιαστική καθυστέρηση και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Αυτά σχετικά με την ψηφιακή οικονομία. Εγώ πιστεύω ότι η καινοτομία πράγματι δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης. Δεν είναι ότι δημιουργεί μόνο έχει καταστρεφικές συνέπειες, κάθε άλλο. Εγώ πιστεύω ότι η καινοτομία συνεπάγεται πολλές ευκαιρίες. Ο τουρισμός μπορεί να διευρυνθεί, μπορεί να διαφοροποιηθεί, να προσφέρει και άλλα πράγματα. Τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ιταλία έχω βιώσει την ανάπτυξη την επέκταση του τουριστικού τομέα. Ως εκ τούτου ε, θεωρώ ότι πραγματικά μπορούν να προκύψουν και νέες δεξιότητες. Τέλος, και ένας φόβος. Ένας φόβος που προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Από τη μια έχουμε πολλές ευκαιρίες, ε, γνωρίζουμε ότι οι αριθμοί συνεχώς ε, θα βελτιώνονται. Πρέπει όμως σε αυτούς τους τουρίστες να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατόν, η εμπειρία τους να είναι αξέχαστη, κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ανοιχτούμε και εμείς για να γνωρίσουμε και τον κόσμο εκτός της Ευρώπης. Δεν θέλουν όλοι μια ιστορική και πολιτιστική εμπειρία. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θέλουν να κάνουν ψώνια, shopping. Και αυτοί λοιπόν αντί ε, να πάνε σε εκκλησίες θέλουν να πάνε σε ένα ε, mall, σε ένα shopping center. Να τα γνωρίζουμε όλα αυτά γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζήτηση και θα μπορούμε να φιλοξενούμε όλο και περισσότερους ε, τουρίστες στην Ευρώπη και να αποδίδουμε όλο και περισσότερα έσοδα στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μοιραστήκατε μαζί μας αυτή την καθημερινότητα του επιχειρηματία που είναι πολύ σημαντική, είναι πολύτιμη για μας. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, επόμενο μιλτή από το Τυρόλο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι με θέματα τουρισμού ε, και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο επιστήμης. Ε, διαπιστώσαμε λοιπόν το πόσο σημαντική είναι η ψηφιοποίηση για την ε, ε, επιστήμη, την έρευνα κυρίως ε, και για την τουριστική ανάπτυξη. Και αυτό τον έφερε σήμερα και η Επίτροπος. Ε, αυτό το είχε εξάλλου επισημάνει και ο προκάτοχός της, ο κύριος Ότιγκερ. Είχε πει ότι ο τουρισμός θα πρέπει να είναι ένας στόχος που να στοχεύουμε στον τουρισμό. Ο υπουργό, ο κύριος Υπουργό από τον τουρισμό από την Ρουμανία ανέφερε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρόσβαση, στην ψηφιοποίηση, αν τα προγράμματα είναι τόσο περίπλοκα που να μην υπάρχει κανένας που να μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνος του και να χρειάζεται συμβούλους. Χρειαζόμαστε την απλούστευση. Απλούστευση των διαδικασιών αλλά και των εργαλείων ενίσχυσης. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι νέες επενδύσεις, χρειαζόμαστε την καινοτομία. Νομίζω ότι τα έχουμε συζητήσει αυτά. Χρειαζόμαστε ε, την χρηματοδότηση, αν θέλετε, και μέσω του προγράμματος ΕΦΣΥ. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ε, μια νέα γραμμή στον προεπιλογισμό, Η Επιτροπή των Περιφερειών πέρυσι το θέμα του τουρισμού ε, η Επιτροπή επικαιροποίησε αυτό το θέμα, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο κύριος Ταγιάννη μας στήριξε ανεπιφύλακτα και ξέρω πολύ καλά ότι ο κύριος Ταγιάννη όταν ήταν επίτροπος ε, είχε ε, ταχθεί ανεπιφύλακτα υπέρ της στήριξη του τουρισμού. Γι' αυτό και εγώ ευχαριστώ θερμά σήμερα για την εκδήλωση. Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή που ασχολείται με θέματα τουρισμού και μεταφορών. Βεβαίως, στο πλαίσιο της ε, ψηφιοποίηση θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσει δεν πρέπει να εξαρτώνται από μονοπόλια ε, και ούτε από διεθνείς πύλες κρατήσεων. Ε, παρακαλώ λοιπόν την κυρία Επίτροπο να το προσέξει αυτό το θέμα. Τελικά να μην καταλήξουμε σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού από την περιοχή των Άλπαιων γνωρίζω ότι έχουν κατατεθεί αρκετές διαμαρτυρίες. Ε, διαφήμιση και η διαφήμιση που είχε κάνει παλαιότερα ο κύριος Ταγιάννη ε, για ταξίδια εκτός Ευρώπης. Ε, αυτά να επανέλθουν η υπηρεσία εξωτικής δράσης, ε, εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να μεριμνά μόνο για διπλωματικές σχέσεις, αλλά να έχει και μία πλατφόρμα για ευαισθητοποίηση σε θέματα τουρισμού. Ένα πράγμα πρέπει να πούμε ότι ο τουρισμός ε, αναμφίβολα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ε, ευρωπαϊκή συνείδηση. Και ε, τον τουρισμό δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο κάτω από καθαρά οικονομικό πρίσμα. Να πω και πρακτικά παραδείγματα. Πρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να προσφέρουμε κίνητρα. Κίνητρα να γνωρίσουν την Ευρώπη των πολιτισμών του χρόνου έχουμε την χρονιά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πώς θα το βλέπατε να έχουμε μια ευρωπαϊκή κάρτα, κάρτα του Ευρωπαίου πολίτη. Αυτό με τη μορφή την πολιτική, ε, την πειραματική σε διάφορες περιοχές. Υπάρχουν πολλοί που προσφέρθηκαν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα. Και μια άλλη δυνατότητα θα ήταν να Έχουμε και ένα GPS φιλικό προς το χρήστη, έτσι ώστε ο Ευρωπαίος πολίτης να αποκτά με μεγάλη ταχύτητα πληροφορίες που αφορούν σε υπηρεσίες ε, υγείας, ε, διπλωματικές υπηρεσίες προξενία. Υπάρχουν πρακτικά ε, παραδείγματα. Εγώ τήρησα το χρόνο που μου είχατε προβλέψει για μένα και ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Σας ευχαριστώ που κρατήσατε, που μείνατε εντός χρονικών όριων. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να αφήσω χρόνο για τη συζήτηση και έχουμε άλλους τέσσερις ομιλητές. Παρακαλώ, μην ξεπερνάτε το χρόνο που σας έχει δοθεί. Ο κύριος Βεν Λάριβακ έχει το λόγο. Στο συγγνώμη αν δεν ε, πρόφερα καλά το όνομά σας. Είναι αντιπρόεδρος του, του Αμαντέους, ε, του ομίλου Αμαντέους για την τεχνολογία των πληροφοριών, για τις ε, ε υποθέσεις της βιομηχανίας και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνατε το λόγο. Το δίκτυο Αδαμαντέους χαίρεται που είναι εδώ. Στοχεύουμε σε μια πανευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό. Μου ζητήσατε να έρθω εδώ και να μιλήσω κυρίως για τις ψηφιακές πλατφόρμες Ίσως γιατί το Αμαντέο το οποίο εκπροσωπώ, είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα και μάλιστα ευρωπαϊκή. Γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε λόγω της απορρίθμισης του κλάδου της αεροπλοείας στην Ευρώπη πριν από 30 χρόνια. Κλείνουμε 30 χρόνια τον επόμενο μήνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε την πρόβλεψη, την πρόνοια και τη σοφία τότε να διασφαλέσει ότι θα υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας για να αποφευθεί η δεσπόζουσα θέση ορισμένων επιχειρήσεων εν ώψη της απορρίθμισης. Προέβλεψε λοιπόν ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν και οι πλατφόρμες για να είναι ουδέτερες με διαφάνεια, για να διασφαλίζουν το δίκαιο ανταγωνισμό, τον θεμητό ανταγωνισμό, να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν πραγματικές επιλογές, αληθινές επιλογές όταν θα συνέκριναν τις προσφορές που θα προέκυπταν εντός συστήματος. Έκτοτε το Μαντέους αναπτύχθηκε, εξελίχθηκε, επεκτάθηκε. Είμαστε μια ψηφιακή επιχείρηση, ο μεγαλύτερος πάροχος ε, τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών στον κλάδο του τουρισμού παγκοσμίας. Είναι μια ιστορία επιτυχίας ή αν θέλετε ευρωπαϊκή ιστορία πρωταθλήματος, πρωταθλητών. Αυτό δείχνει ότι η αν θελετε ευρωπαικη ιστορια πρωταθληματος πρωταθλητων αυτο δειχνει οτι οι εταιρείε τεχνολογίας μπορούν να ανθούν σε ένα σωστό πλαίσιο που είναι ρυθμισμένο και επιτυχάνει το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ του ελεύθερου επιχειρήν από τη μία και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από την άλλη. Ε, με βάση τη διαφάνεια, τις αληθινές επιλογές, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια. Επομένως, εμείς στο κλάδο της αεροπλοείας υποκείμεθα σε συγκεκριμένη νομοθεσία που είναι πολύ συγκεκριμένη, ως προς, για παράδειγμα, την κατάταξη των πτήσεων που βλέπει ο καταναλωτής όταν τις βλέπει συγκριτικά, και η επιτυχημένη ιστορία της απελευθέρωσης και της απορρίθμισης της αεροπλοείας στην Ευρώπη έχει πολλά μαθήματα να κομίσει, πάρα πολλές εμπειρίες να συνεισφέρει στο διάλογο, τον ευρύτερο διάλογο, έτσι ώστε οι αρχές αυτές να εφαρμοστούν και σε άλλους κλάδους. Όταν κανείς παίρνει απόσταση, κοιτάζει τη συνολική εικόνα, έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει ε, δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση ε, υπάρχει προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Γίνεται λόγος για τον τουρισμό, αλλά να μην ξεχνούμε ότι μιλούμε και για επιχειρήσεις. Ε, για επιχειρηματικά ταξίδια, αλλά και για ατομικά ταξίδια. τα επιχειρηματικά ταξίδια υποτίθεται ότι είναι και ο λόγος ουσιαστικά και είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να ξοδεύουμε ατομικά ταξιδεύοντας στη συνέχεια στον προσωπικό μας χρόνο. Και αυτό πρέπει κανείς να το έχει υπόψη του. Ε, μιλούμε για την Ευρώπη ως προορισμός διακοπών. Ωστόσο, το 85% των επισκεπτών αυτών είναι εντός Ευρώπης. Άρα, μιλούμε για τον Ευρωπαίο καταναλωτή, για τον Ευρωπαίο πολίτη. Μιλούμε για πολιτικές και προγράμματα και πώς αυτά θα θεσμοθετηθούν που θα βελτιώσουν τη ζωή όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και άρα Μιλούμε για την προσβασιμότητα με την πολύ ευρία έννοια αυτής της λέξης. Προσβασιμότητα, πρόσβαση σε μία αγορά για να δρέψει κανείς τα ωφέλη αυτής της αγοράς. Είτε είναι πάροχος, είτε είναι ε, παίκτης της αγοράς που συνδέει ε, άλλους εταίρους μεταξύ τους. Θα ε, παρουσιάσουμε μία λευκή βίβλο την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε τα άτομα με, αναπηρία, ε, με αναπηρίες να έχουν καλύτερη πρόσβαση Μιλούμε λοιπόν για πρόσβαση σε μια αγορά για τα δικαιώματα των παικτών στην αγορά, είτε πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για π.χ. καταναλωτές με απαιτήσει στον τομέα των αναπηριών και ούτω καθεξής. Χαιρόμαστε που διεξάγουμε αυτό το διάλογο με εσά, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς από τους παριστάμενους και με μεγάλη χαρά θα συμμετάσχουμε και στη συνέχεια αυτής της ε, διαδικασίας. Ευχαριστώ η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σβέν Λάιρβακ γιατί αναφερθήκατε και στα επιχειρηματικά ταξίδια και πράγματι συγχαρητήρια. Το Αμαντέους είναι πρωταθλητής, Ευρωπαίος πρωταθλητής που δείχνει ότι η Ευρώπη μπορεί. Στη τελευταία ολομέλεια του Στρασβούργου ψηφίσαμε το ε, νομοθέτημα για την προσβασιμότητα είναι νομοθεσία για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, πρόσβασης και για άτομα με αναπηρίες. Και αυτό είναι ένα σημαντικότατο βήμα προς τα εμπρός. Με πολύ μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο στον κύριο Χαβιέ Σελντράν, Περιφερειακό Υπουργό Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος της ε, Περιφέρειας της Μούρθιας στην Ισπανία. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσω την άποψή μας για την ψηφιακή μετάβαση του κλάδου του τουρισμού. Η Μούρθια είναι μια μικρή αλλά πολύ δυναμική σφίζουσα περιοχή της Ισπανίας στη Μεσόγειο με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους πληθυσμού. Έχουμε ένα πολύ έντονο τουριστικό κλάδο. Το 2016 δεχθήκαμε 5,3 εκατομμύρια τουρίστες και 39 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Οι τουρίστες συμβάλλουν στο περιφερειακό μας ΑΕΠ κατά 11%, αύξηση 5% το 2016. Σε αυτό το πλαίσιο η περιφέρεια της Μούρθια έχει απο... θεωρεί ότι η βιομηχανία φιλοξενίας και καταλημάτων ε, είναι κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και γι' αυτό σχεδιάσαμε τη στρατηγική 2015-2019 για τον τουρισμό και καθορίσαμε τα πρώτα βήματα για να έχουμε μια δομική ανασυγκρότηση, μια δομική αλλαγή ε, στο τουριστικό προϊόν και να καλύψουμε τις ανάγκες του ψηφιακού τουρίστα. Όλες οι στρατηγικές και οι δράσεις βάσει του στρατηγικού σχεδίου εστιάζονται στο να ε, ικανοποιήσουμε τα νέα προαπαιτούμενα του εφιούς ταξιδιώτη δηλαδή να έχουμε μια προσφορά customized, προσαρμοσμένη στις απαιτήσει και στις εκάστοτε ανάγκες. Εστιάζουμε την προσοχή μας σε βασικά προϊόντα που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, που μπορούν να ενισχύσουν και να αυξήσουν τα εισοδήματα και τα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και που μπορούν να προσελκύσουν νέες επενδύσεις σε βιώσιμα αηφόρα επενδυτικά σχέδια τι σημαίνει να προσαρμοστούμε στον ε, ε, έξυπνο ή ευφυή ταξιδιώτη. Άρα να είμαστε εμείς σε πρωτοπόροι σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Να καταρτιστούμε καλύτερα στις ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό είναι ε, προαπαιτούμενο για να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα. Τα big data, οι έξυπνες εφαρμογές, το ψηφιακό marketing, η συγκέντρωση πληροφοριών για τις επιχειρηματικές συνήθειες, τα μέσα κοινωνικής κοινωνικής δικτύωσης είναι όλα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να ενισχύσουμε την τουριστική μας στρατηγική και υπάρχουν διάφορα καλά περιαδείγματα που δείχνουν πώς ένα ηλεκτρονικό προϊόν μπορεί να αποτελέσει μια ιστορία επιτυχίας και πώς ε, μπορούν να συστρατευτούν όλοι και το ευρωπαϊκό και το κρατικό και το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. Η Καραμπάκα Ντελακρούθ είναι μια μικρή πόλη στη Μούρθια, μία από τις πέντε ιερές πόλεις του κόσμου. Τρεις από αυτές βρίσκονται στην ε, Ισπανία. Είναι βασικός προορισμός για προσκυνητές, για ανθρώπους που θέλουν να ε, πάνε σε μέρη που είναι ευχάριστα αλλά και που θα τροφοδοτούν το πνεύμα και τη σκέψη. Αξιοποιούνται όλες οι τεχνολογικές δυνατότητες που παρέχει η περιφέρεια Έχουμε ένα σύστημα το ΆΡΠΑ για άμεσες κρατήσεις για τους προσκυνητές, ειδικέ εφαρμογές για τους προσκυνητές. Έχουμε την πλατφόρμα ε, την ψηφιακή Nexo με βάση τα big data για να καταλάβουμε καλύτερα τις συνήθειες των προσκυνητών. Έχουμε την Orient, μια άλλη πλατφόρμα για να πουλήσουμε δραστηριότητες και ε, πακέτα στους προσκυνητές. Έχουμε δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα ε, θέση σε εμπορία και θέσεις στην αγορά των τουριστικών προϊόντων των επιχειρήσεων που λέγεται Ερμής η πλατφόρμα αυτή και ε, είναι δωρεάν η χρήση στους τελικούς χρήστες και αλλά και σε άλλους παρόχους. Ήταν το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής καλυψούς, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ένα σημαντικό βήμα για ε, τις ανταλλαγές μεταξύ διαφόρων ψηφιακών πλατφορμών. Τέλος, θέλω να τονίσω την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, όπως πρότεινε και ο πρόεδρος Ταγιάννη. Ο Περιφερειάρχης της Μούρθια στηρίζει την επιστολή που απέστη απεστάλει στον πρόεδρο Γιούνκερ τον Ιούλιο, όπου ζητάτε να συμπεριληφθεί αυτό στο νέο πρόγραμμα δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2018 και μετά. Είναι κοινέ οι προκλήσει και πρέπει με εγκάρσιο τρόπο να τι αντιμετωπίζουμε σε όλε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και με προοπτικέ μακροπρόθεσμε. Να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να εξοπλίσουν πλήρω το δυναμικό τη ψηφιακή οικονομία, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να του δώσουμε αρκετέ ευκαιρίε να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, να να δώσουμε χρηματοπιστωτικά και χρηματοοικονομικά εργαλεία για να αναπτύξουν στρατηγικές, να ανταποκριθούν στις ψηφιακές προκλήσεις. Πρέπει να στηρίξουμε το, ε, την πύλη για τις επενδύσεις, το hub ε, και όλες αυτές τις ε, ηλεκτρονικές δράσεις που ενισχύουν τις δεξιότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Σελτράν. Προτείνετε να συμπεριληφθούν κάποια στοιχεία στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαντάζομαι ε, τα κατέγραψε λεπτομεριακά όλα αυτά η κυρία Επίτροπος. Περνάμε στον κύριο Φερχόφεν, που είναι διευθυντής των εταιρικών υπηρεσιών και διευθυντής ΕΜΕΑ της Booking.com. Παρακαλώ τέσσερα λεπτά, όχι παραπάνω. Σα ευχαριστούμε για την πρόσκληση για να πούμε πώ μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερου πελάτε στην Ευρώπη. Αυτό είναι το βασικό θέμα και ίσω αυτό θα πρέπει πρώτα να αναλύσουμε πριν να περάσουμε στι λεπτομέρειε τη φορολογία και ποιο παίρνει τμήμα του μεριδίου, τμήμα τη Πίτα. Να δούμε πώ θα αυξήσουμε, θα επεκτείνουμε την πίτα. Είμαστε από τι βασικέ πλατφόρμε που διαδραματίζουν ρόλο κλειδί. Ε, ε, το 1996 ιδρυθήκαμε στην Ολλανδία και έχουμε την εταιρική μας έδρα στο Άμστερνταμ. Απασχολούμε 5.000 ανθρώπους, περίπου από 100 εθνικότητε και από ε, τον ξενοδοχειακό κλάδο, ε, από, τις, από διάφορες επιστήμες, τεχνολογία και πληροφορίε, αλλά πολλούς και από το ξενοδοχειακό κλάδο και θέλουμε να εξυπηρετήσουμε του εταίρους μα. Γι' αυτό και έχουμε διάφορα σεμινάρια για τεχνολογίες πληροφορίες. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια γίναμε το βασικό, η βασική ιστοσελίδα για, τις, ε, για τη στέγαση τουριστών ε, και παρά το, την περιαγωγή ε, είδαμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις μετακινήσεις και να μειώσουμε τους, τους, τις τριβές στην προσφορά της πληροφορίας. Και μάλιστα ε, η προσφορά υπηρεσιών με την καλύτερη τιμή στον πελάτη, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θέλουμε να προσφέρουμε στον πελάτη με τους εταίρους μας. Είμαστε η εκδοχή της 20 του 21ου αιώνα του καταλόγου ταξιδιών. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε σε ένα ενίο μέρο όλε τι προσφορέ με διαφανή και αξιόπιστο περιβάλλον, ώστε να μπορούν να βρουν προορισμού παντού στον κόσμο οι πελάτε, ανάλογα με τα γούστα του και τι προτιμήσει του διανυκτερεύσεις, ε, σε καταλήμματα, σε ξενοδοχεία με όλους τους όρους και συνθήκες ανάλογα με τις τιμές που διαθέτουν οι πελάτες. Και μάλιστα η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν. Ε, και η πληρωμή γίνεται μόνο όταν γίνεται κράτηση ε, και μάλιστα η φορολογία των, της προμήθειας που κρατούμε γίνεται στις κάτω χώρες και όλα τα υπόλοιπα που δεν αφορούν την προμήθεια παραμένουν και φορολογούνται στη χώρα προορισμού. Η πλατφόρμα αυτή, το Booking.com, δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες και για τους εταίρους και για τους ε, καταναλωτές. Έχουμε 1,4 εκατομμύρια καταλήμματα, 26 ε, ε, δωμάτια, εκατομμύρια δωμάτια συνολικά και βλέπουμε τα πλεονεκτήματα για τους πολίτες. Καταρχήν, είμαστε εταίροι τεχνολογίας για τα, για τα ξενοδοχεία, κυρίως τα μικρά, τα ανεξάρτητα, που είναι τρία τέταρτα των κρατήσεων. ε, ξενοδοχεία, ξενώνες, καταλήματα. Είμαστε η πύλη για τη διεύρυνση των, ε, της βάσης ε, πελατών με χαμηλό κόστος, πολύ χαμηλότερο από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης, ε, φέρουμε πελάτε στα ξενοδοχεία, αυξάνοντα την πληρότητά του. Πελάτε που δεν θα μπορούσαν να προσελκύσουν μόνο του τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα, γιατί προέρχονται από κάθε περιοχή του κόσμου, κυρίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Όλη μου τη ζωή απασχολήθηκα στο ξεροθοχειακό κλάδο. Τότε για να ανοίξει κανεί ε, μια τέτοια επιχείρηση ε, ε, πρέπει να περάσουν μήνε για να επιτυχεί μεγάλη πληρότητα. Χάρη στι πλατφόρμε σαν τη δική μα, τέτοια καταλήματα ανοίγουν αμέσω και μπορούν να εξασφαλίσουν πληρότητα μέσα σε λίγε μέρε ή εβδομάδε και να γίνουν προσοδοφόρε επιχειρήσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Επίση, εξασφαλίσουμε μετάφραση 43 γλώσσες ε, των προσφορών, 24 ώρες, 24 πρόσβαση και οι ιδιοκτήτες των καταλημάτων μπορούν να αποφασίσουν τι, πόσα δωμάτια διαθέτουν, σε τι ποσοστό και με τι πολιτική ακύρωση. Και όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν όλες αυτές τις συνθήκες ανα πάσα στιγμή μέσω του εξωτερικού δικτύου. Επίσης, ένας πελάτης από την Κίνα μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει με ένα πορτογαλικό κατάλημα χάρη στη μετάφραση που εξασφαλίζουμε μία από τις προσφορές στους πελάτες. Επίσης και για τους καταναλωτές είναι πολύ σημαντική εύκολη πρόσβαση. Ε, εύκολη πρόσβαση φιλική προς το χρήση, χρήστη που μπορεί να κάνει σύγκριση των τιμών, οπότε μπορεί να ταξιδέψει πολύ πιο άφοβα συγκρίνοντας ε, τις προσφορές ε, στις διάφορες πλατφόρμες. Έχουμε ε, άπειρες κριτικές που διευκολύνουν τους πελάτες να κάνουν τις επιλογές τους. Έτσι κάνουμε πραγματικότητα την ενιαία αγορά και επικεντρωνόμαστε στις ευκαιρίες για τους καταναλωτές και όχι στους φόβους της ψηφιοποίησης. Καταπολεμούμε την αυξανόμενη, τον αυξανόμενο κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς, να, προσπαθώντας να άρουμε τα εμπόδια που την υπονομεύουν θα πρέπει να μας θεωρήσετε ως εταίρους και όχι τους εχθρούς της συμβατικής τουριστικής δραστηριότητας. Είμαστε το μέλλον και θα βοηθήσουμε τον τουρισμό προσελκύοντας περισσότερους πελάτες, περισσότερους τουρίστες στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φεχόιερ από την booking.com. Περνάμε τώρα στον τελευταίο μας ομιλητή, τον Λουίτζι Γκαμπαρντέλα, που είναι πρόεδρος της εταιρείας China EU. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ, τα υπερβείτε. Σας ευχαριστώ. Δεν Και... Ευχαριστώ τον κύριο Ταγιάννη που οργάνωσε αυτή την τόσο σημαντική σημερινή συνάντηση. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δύο λέξεις κλειδί για τον ε, τουρισμό, το μέλλον του τουρισμού στην Ευρώπη. Οι λέξεις ψηφιακό και οι λέξεις Κίνα. Όπως ανέφερε προηγουμένως και η Επίτροπος, η κυρία Γκάμπριελ, ε, η ψηφιακή εξέλιξη είναι πολύ σημαντική για τον τουρισμό. Και το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι το εξή. Ε, το ψηφιακό στοιχείο, ε, γενικά η ψηφιακή τεχνολογία, αλλάζει όλο το θέμα του τουρισμού και προσφέρει άλλε δυνατότητε στον τουρίστα. Του δίνει τη δυνατότητα να έχει και μία τελείω διαφορετική εμπειρία. Το δεύτερο όμω που είναι πιο σημαντικό είναι ότι χάρη των big data που αναφέρθηκαν, των μέσων κοινωνική δικτύωση και τι τεχνικέ ε, τη τεχνητή νοημοσύνη, σήμερα μπορεί πλέον κανεί να προβλέψει ε, το πότε θέλει κάποιος να πάει διακοπές. Το πότε θα πάει και πού ενδεχομένως θα θελήσει να πάει. Αυτό είναι το ψηφιακό μάρκετινγκ. Εγώ πιστεύω όμως ότι η ερώτηση που πρέπει να βάλουμε ως Ευρωπαίοι είναι κατά πόσον ο ευρωπαϊκός τουρισμός είναι έτοιμος να δεχτεί αυτή την αλλαγή, αυτή την ψηφιακή επανάσταση με τα 5G θα ξεκινήσουν βεβαίως και πολλές άλλες δυνατότητες. Ε, η δεύτερη λέξη κλειδί είναι, όπως είπα, η Κίνα. Γιατί, διότι το δυναμικό είναι τεράστιο. Στο Νταβός, ε, στο τελευταίο Νταβός, ακούσαμε ότι η Κίνα προτίθεται να στείλει 700 εκατομμύρια Κινέζους τουρίστες κατά τα αμέσω επόμενα έτη. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Κινέζοι τουρίστες στην Ευρώπη είναι μόνο 10 εκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν τι τεράστιες δυνατότητες υπάρχουν σε σχέση με αυτή την αγορά. Το Σίτριπ το κινέζικο που είναι ανταγωνιστής ε, του Booking ε, έχει περίπου 300 εκατομμύρια εισιτήρια το χρόνο για να έχετε μια ιδέα για το τι πράγμα μιλάμε. Μπροστά λοιπόν σε όλες αυτές τις ευκαιρίες που προσφέρονται θα ήθελα να κάνω μια πρόταση και εκμεταλλεύομαι βέβαια και την παρουσία της Επιτρόπου που έχει μια, ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο για την Ευρώπη και για όλους μας. Η πρόταση αυτή είναι η εξή. Η επόμενη χρονιά θα είναι η χρονιά τουρισμού ανάμεσα στην Ευρώπη και την Κίνα. Νομίζω ε, θα ξεκινήσει, τα γέννη θα τα έχουμε στις 19 Ιανουαρίου ε, στην Βενετία. Ε, πρέπει τώρα λιγάκι να, να κάνουμε κάποια προγράμματα ως ε, Ευρωπαίοι. Εγώ νομίζω ότι και με την βοήθεια της Επιτρόπου θα έπρεπε να οργανώσουμε στη Βενετία μια στρογγυλή τράπεζα που θα συμμετέχει η ψηφιακή οικονομία, οι Κινέζοι και οι Ευρωπαίοι και όλοι μαζί να επεξεργαστούν κάποιες προτάσεις που θα επιτρέψουν να φτάσει τουλάχιστον να φτάσουν τα 20 εκατομμύρια οι Κινέζοι τουρίστες στην Ευρώπη ε, το 2020 και να αυξηθούν και οι δαπάνες αυτών των τουριστών. Δηλαδή να έχουμε ένα Κινέζο τουρίστα που θα δαπανά περισσότερα χρήματα στην Ευρώπη. Γιατί ε, μερικές φορές μιλάμε για την Κίνα αλλά ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι και ήπειρος. Ως εκ τούτου ε, και σε σχέση με τον τουρισμό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα αυτήν την αγορά. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ. Νομίζω έμεινα στα τέσσερα λεπτά, έτσι δεν είναι. Τέλεια, πράγματι. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε αυτές τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η Κίνα για την Ευρώπη. Και τώρα θα ήθελα όλοι να καταχειροκροτήσουμε το καταπληκτικό μας πάνελ των καλεσμένων και να περάσουμε στη συζήτηση. Ε, να ακούσουμε τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, αλλά γρήγορα παρακαλώ. I'm sure this panel has been very inspiring for many. Φαντάζομαι ότι θα σας ενέπνευσε αυτό το πάνελ, παρόλο που είναι προχωρημένη η ώρα, πήγε αυτά το απόγευμα. Δεν, φαντα... Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μετά αυτά που ακούσαμε από την Booking.com, ε, κανένας ε, δεν σκέφτηκε να υποβάλει ερωτήσεις. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Εγώ μαζί με το επιτελείο μου έχουμε τη χαρά να ταξιδεύουμε παντού στον κόσμο και να μιλούμε με εκπροσώπους και ενδιαφερομένων και του κλάδου και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως κοινότητα είναι τεράστιες ε, γιατί είναι πολλές οι ευκαιρίες, αλλά και οι προκλήσεις είναι εξίσου σοβαρές. Γιατί δημιουργούνται πια νέες ανάγκες ε, συνεργασίας δημόσιο και ιδιωτικού κλάδου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα αναλύοντας, ε, αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις. Είναι νέες οι προκλήσεις και θα πρέπει να αλλάξουν και τα μοντέλα των σχέσεών μας. Γιατί από τη σκοπιά των ενδιαφερομένων ε, δεν πρέπει να σταματούμε να... Ίσως πρέπει να σταματούμε να περιμένουμε από την Ευρώπη και να κάνουμε και εμείς κάτι για την Ευρώπη και να συμβάλλουμε και εμείς στην κοινή μας πρόοδο. Ε, σίγουρα εκτιμούμε ιδιαίτερο στο σχόλιο σας και εγώ και η Επίτροπος Μαρία Γκαμπριέλ και φαντάζομαι και οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα σχόλια ή ερωτήσεις. Uh, Έχω να ρωτήσεις, ναι. Μία ερώτηση έχω να υποβάλω, η οποία ερώτηση έχει σχέση ε, με την ανανέωση, την καινοτομία και σε σχέση με τις ε, πλατφόρμες πληρωμής. Νομίζω ότι ε, γίνονται με μεγάλη ταχύτητα οι πληρωμές και αυτό ε, μπορεί να δημιουργήσει όμως και πάρα πολλά προβλήματα. Ο δικός μας ο κλάδος ε, ε, πρέπει να διατηρήσει και να διαφυλάξει και την ιδιωτικότητα. Αυτό είναι σαφής υποχρέωση για μας και για τον κλάδο μας. Ε, βεβαίως, πρέπει, όπως σας είπα, να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, αλλά αυτό σημαίνει και ότι θα υπάρξουν και μεγάλες αλλαγές στις πλατφόρμες. Σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί επιβάλλεται τόσο υψηλά πρόστιμα. Αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω να υποβάλω. Σε ποιον την υποβάλλετε, σε εσά. Ε, ε, Ευχαριστώ. Um, uh, το είχα πει και προηγουμένως το θέμα του κανονισμού για την ε, ηλεκτρονική ιδιωτική σφαίρα, το e-privacy και μάλιστα αύριο στην, αγορά εσωτερι... στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και προστασία του Καταναλωτή θα ψηφίσουμε επί της νομοθετικής πρότασης για το e-privacy, την ιδιωτικότητα στο, στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να μπορούμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα σε μια οικονομία που είναι προσανατολισμένη προς τα δεδομένα, ακόμη και στον τουριστικό κλάδο. Μέχρι στιγμής ε, ε, προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ Τη ιδιωτικότητα και της ανάγκης ανταλλαγή δεδομένων στο τουριστικό τομέα. Ακόμη δεν τη βρήκαμε αυτή την ισορροπία, γιατί έχουμε τη διαφήμιση, την επιλογή του καταναλωτή, την ψυχαγωγία του καταναλωτή και τη δυνατότητα πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αναπτύξουν επιγραμμικά τις υπηρεσίες τους. Άλλος κανείς θέλει να προσθέσει κάτι. Any more questions or comments? Άλλα σχόλια ή ερωτήσεις. Νόρμα ε, Κλάρκσον, εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Ξεναγών. Ε, το επάγγελμα του ξεναγού βρίσκεται υπό εξαφάνιση. Έχουμε σε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό ε, τον ορισμό ε, έχουμε τώρα τις δωρεάν αυτές ξεναγήσεις που δεν είναι και πολύ δωρεάν γιατί ο καταναλωτής ε, ε περιμένει από τον καταναλωτή ένα φιλοδόρημα στο τέλος ε, και πρόκειται για ενειδίκευτους ξεναγούς δεν μπορούν να διαχειριστούν ομάδες, καταστρέφουν πολιτιστικά αξιοθέατα, εξοργίζουν τους ντόπιου και δίνουν και ανακριβείς πληροφορίες. Αυτή είναι απειλή για τους επαγγελματίες ξεναγούς. Μερικές φορές είναι άσχετη και με τη χώρα στην οποία ξεναγούν τα γκρουπ. Πώς βλέπετε λοιπόν ε, την εξασφάλιση συνθήκων θεμητού ανταγωνισμού για το επάγγελμα των ξεναγών. Θέλει κανείς απαντήσει. Ο κύριος Ντάντι. Επανειλημμένα. Είχαμε αυτή τη συζήτηση σχετικά με τους ξεναγούς. Όπως είπατε, βρισκόμαστε πλέον σε μια φάση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει ένα κείμενο στα κράτη-μέλη σχετικά με την αναγνώριση κάποιων επαγγελμάτων, μεταξύ αυτών και των ε, ξεναγών. Ε, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ένα ισορροπημένο, εξορροπημένο κείμενο έτσι ώστε τα κράτη ε, να μπορούν να εγγυούνται ότι δεν θα υπάρχουν καταχρήσεις σε, αυτό το επάγγελμα το οποίο ε, επάγγελμα και όσοι ασκούν αυτό το επάγγελμα είναι σαφές ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να το ασκούν, να έχουν τι απαραίτητες γνώσεις. Όσον αφορά τη συνεργατική οικονομία, νομίζω είναι απόλυτα σαφές. Δεν ξέρω ε, πόσοι μπορούν να ε, προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Πρόκειται για επαγγελματική φύσεως υπηρεσίες και εμείς ανέκαθεν είχαμε κατά νου μία αρχή ότι οποτεδήποτε πρόκειται για επαγγελματικές υπηρεσίες η προϋπόθεση για το ποιος θα λειτουργεί σε μία ε, ψηφιακή πλατφόρμα και ποιος θα λειτουργεί με παραδοσιακό τρόπο, τα κριτήρια θα πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες που θα δίνουν τη δυνατότητα του σαφούς ε, διαχωρισμού, άρα δηλαδή να μην ε, ισχύουν ειδικέ προϋποθέσεις πέρα από τις ευρωπαϊκές. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό και ε, πιστεύουμε ότι θα γίνει και το πρώτο βήμα για την αναγνώριση του επαγγέλματος για να καλύπτονται και οι ξεναγοί. Σε ευχαριστούμε Νικόλα. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, να ολοκληρώσω τη συζήτηση συνοψίζοντα κάποια θέματα που έχουμε επιτάπητος και μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Καταρχήν, είμαστε πλήρω προσιλωμένοι στην ανάγκη ολοκλήρωση τη ενιαία ψηφιακή αγορά. για να καταργήσουμε τον κατακαιρματισμό, να διευκολύνουμε τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και να εναρμονίσουμε του κανόνε για να μειώσουμε το κόστο και τη γραφειοκρατία, κυρίω για τι μικρομεσαίες αλλά και για τι μεγάλε επιχειρήσει. Τώρα επεξεργαζόμαστε το πακέτο για τι υπηρεσίε. και όταν βλέπω τον κατάλογο με του τομεί που καλύπτονται από την ηλεκτρονική κάρτα, το e-card, περιλαμβάνονται και τα ταξιδιωτικά πρακτορία, οι tour operators και άλλες συναφείς δραστηριότητες με τον τουρισμό. Οπότε πολύ ευχαρίστω να έχουμε διάλογο και μαζί σας για το θέμα αυτό. Είμαι και συγγήτρια του κανονισμού για το ΕΛΚ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι εργάζονται άοκνα προκειμένου να καταλήξουμε σε καλή πρόταση. Ξέρω πόσο σημαντικός είναι και ο κανονισμός για την ε, ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο. Πολύ αναφερθήκατε στην ανάγκη που έχει επιλογή, ψυχαγωγία και προστασία του καταναλωτή. Και οι νέοι τρόποι φροντίδας του πελάτη που έχουν αναπτύξει ή φέρει ε, οι νέες πλατφόρμες. Και μάλιστα έχουμε αναθεωρήσει ε, το νέο πακέτο της ε, ταξιδιωτικής οδηγίας του 2015 που θα τεθεί σε ισχύ και που θα αυξήσει την προστασία του καταναλωτή στην ψηφιακή εποχή. Η Μαρία αναφέρθηκε στο γεωγραφικό αποκλεισμό. Δεν θα είναι πιο δυνατό να προσφέρονται διαφορετικές προσφορές σε διαφορετικές τιμές στους καταναλωτές ανάλογα με το που βρίσκονται. Ήδη ε, έχουμε καταργήσει τα τέλη περιαγωγής και στο νέο πακέτο για των οδηγιών για τα ταξίδια που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2018 θα ληφθούν υπόψη πολλές από τις ρηξικέλεθες αλλαγές που επέφερε η ψηφιακή επανάσταση και στα ταξίδια και στους καταναλωτές. Και σίγουρα η αξιοπιστία είναι το νέο νόμισμα. Είναι σημαντικό τμήμα και της προστασίας του καταναλωτή. Γιατί ο καθένας μπορεί να βαθμολογεί και να αξιολογεί τις υπηρεσίες που έχει λάβει. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που εξετάσαμε σήμερα είναι ότι δεν θα πρέπει να μείνει κανένας πίσω, να μην μείνει κανείς αποκλεισμένος και να μην εκδιωχθεί αυτό το μονοπάτι της αλλαγής, αυτό το δρόμο της αλλαγής που είναι ραγδαίος και πολλοί παραδοσιακοί ε, πάροχοι νιώθουν την απειλή της νέας επανάστασης. Γι' αυτό με τη συνεργατική οικονομία, με την αύξηση νέων τελεστών στην αγορά. Δημιουργούνται διαφορετικέ συνθήκε. Εμεί έχουμε δεσμευτεί να εξασφαλίσουμε διαφάνεια και συνθήκε θεμητού ανταγωνισμού για όλου. Φυσικά ε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την αυτοματοποίηση και αυτούς που θα χάσουν τη δουλειά τους, αλλά είμαστε δεσμευμένοι και έχουμε υποσχεθεί ό,τι και να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μην αφήσουμε κανένα πολίτη πίσω. Και μια καινοτόμα επιχείρηση και μια παραδοσιακή επιχείρηση να μπορούν να συνεχίσουν να ε, τις δραστηριότητές τους και να προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα. Και το θέμα των αλγορίθμων επίσης. Πώς εντάσσεται και αυτό το θέμα στο θεμητό ανταγωνισμό. Και αύριο οι κατευθυντήριες γραμμές για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πλατφόρμες θα αναθεωρηθούν επίσης. Και πριν εν είδη αστεισμού ή εν είδη πρόκλησης αναφέρθηκα στην Booking.com. Δεν ήθελα να κατονομάσω ένα μόνο εταίρο, ε, την Booking.com ή το Amadeus ή καμία άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πάντως, όπως είδαμε από τι παρεμβάσεις, είναι πολύ έντονα τα πάθη και όπως είπαν πολλοί, υπάρχουν ουσιαστικέ ανησυχίες και εύλογες ε, ανησυχίε, γιατί πολλοί στην Ευρώπη εξαρτώμαστε από τις μεγάλες αυτές πλατφόρμες και δεν θα ήθελα να προτιμηθεί η μία ή η αλλη αλλά μας περιγράψατε μία καταπληκτική και πανέμορφη εικόνα για την επιχείρησή σας. Όλοι φυσικά γνωρίζουμε την Booking.com, είναι πασίγνωστη ε, στο σελίδα, αλλά υπάρχει το θέμα του θεμετού ανταγωνισμού και της εξάρτησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ είμαι υπέρ των ανοιχτών αγορών, του ανοιχτού διαδικτύου, ε, της οικουμενικής ε, ασφαλούς πρόσβασης για όλους και προσιτής πρόσβασης. Πάντως πραγματικά όλα αυτά τα σχόλια θα τα λάβουμε υπόψη. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τον διάλογο. Χρειαζόμαστε τη δική σας εμπειρογνωμοσύνη, τις εμπειρίες και τα βιώματά σας. Και φυσικά δεν έχουμε την αξίωση να τα επιλύσουμε ή την ελαζονία να τα επιλύσουμε από μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Και τώρα, εκ μέρους του Πρόεδρου Ταγιάννη, σας καλώ όλους σε μια δεξίωση που θα παρασχεθεί στο εστιατόριο των Ευρωβουλευτών, ανοιχτή σε όλους, στο ισόγειο του κτηρίου ΑΣΠΕ, δηλαδή με το που θα βγείτε αριστερά στην πλατφόρμα και κάτω στο ισόγειο. Ευχαριστώ και ας εισπυρώσουμε τις δυνάμεις μας. Καλό σας βράδυ.